Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ακολουθεί η προφορική ερώτηση προς